στις 11.30. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας. Επόμενη σύνοδος της Ορομελίας, την 3η, 10 Δεκεμβρίου 2013, ε, από τις 8.30 μέχρι τις 3, ε, μέχρι τις 2, συγγνώμη, και ξανά ε, το απόγευμα. Όλες οι σημερινές συζητήσεις θα βρίσκονται